λειτουργούν τα μηχανήματα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, πέρασε τη ψηφοφορία. Λειτουργεί, μια χαρά, επομένως μπορούμε να ξεκινήσουμε. Τροπολογία 46, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 47, υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος, άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, πέρασε της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 49 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ήσασταν κατά για το δεύτερο τμήμα, συγγνώμη. Επαλήθευση λοιπόν για το δεύτερο τμήμα. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι ψήφισαν κάποιοι από την ομάδα σας. Δεύτερο τμήμα τη. 49, επαλήθευση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έχετε δίκιο. Δεν ελέγχουμε το πρώτο τμήμα. Τροπολογία 50. Αν θέλετε, Κριστιαν, να περάσουμε όλο μας το πρωί εδώ, μπορούμε να συνεχίσουμε να ψηφίζουμε. 50 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 54 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση της 65, νομίζω εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία.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 Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 87 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση για την 88. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται, 92 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 93 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 94 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 95 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση της 95, άρχεται η ψηφοφορία. Νομίζω εγκρίνεται. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 96 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 98 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση της 98, άρχεται η ψηφοφορία. Νομίζω εγκρίνεται. Ψήφισαν όλοι, πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 99 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 101 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 102 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 103 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 110 σε τρία τμήματα. Πρώτα τμήμα με προφορική τροπολογία 2 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τμήμα 1 υπέρ, κατά, α, συγγνώμη, αυτό καταπίπτει, δεν το ψηφίζουμε. Τμήμα 2 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, πέρας της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 111 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Επαλήθευση της 111, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 113 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 112 υπέρ, κατά, αποχές, Επαλήθευση της 112. Άρχεται η ψηφοφορία. Συγγνώμη, καταπίπτει γιατί εγκρίθηκε η 111. Συγγνώμη, δεν χρειάζεται να επαληθεύσουμε. «114 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 48 καταπίπτει Καταπίπτει και 8. Συμβαστική τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 124. Υπέρ. 124. Υπέρ. Υπέρ. Ξανά. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 14 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 15 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. 136 υπέρ, κατά αποχέ απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 17 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 18 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 145 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση της 145 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται Συμβαστική τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική τροπολογία 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 151 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 20 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση 155, άρχεται ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 156 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 157 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Επαλήθευση της 157, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 158 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 159 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 160 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 161 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 162 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 163 αποσύρθηκε, 164 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 165 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα της 165 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 166 υπέρ, κατά αποχές επαλήθευση της 166 άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 167 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 168 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 161 υπέρ. Κατά αποχές. Επαλήθευση της 169. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 170 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 171 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 172 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 173 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 174 υπέρ. Κατά αποχές επαλήθευση της 174. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 179 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 182 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 28 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 24 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 189 αποσύρεται, 190 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 192 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 191 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 193 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 194 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Επαλήθευση 194, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, πέρας της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 195. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ. Ε, εγκρίνεται. 199 υπέρ αποχές 200 υπέρ κατά αποχές 203 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 203 αρχή της ψηφοφορίας ψήφισαν όλοι τέλος εγκρίνεται 26 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 205 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 207 υπέρ κατά αποχές. Ελέγχουμε την 207. Ψηφίσατε. Κάτι δεν πήγε καλά. Ψηφίζουμε. Συνεχίζει ψηφοφορία επί της 207. Ελέγξτε ότι έχετε ψηφίσει όλοι. Τέλος. Τέλος. Εγκρίνεται. 209 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 210 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβεβαστική 1. Εγκρίνεται. 12 υπέρ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 Κατά. Απόχες. Ελέγχουμε την 21, αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 22, αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε. Εγώ δεν ψήφισα. Τέλος. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 26. Τέλος. Απορρίπτεται 26. 29 συμβαστική υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά αποχές. Ελέγχουμε την 29. Τέλος. Απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος για την 31. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται η 31. 32 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 κατά πίπτη, προφορική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές Έλεγχος. Ελέγχουμε την 38. Τέλος. Εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά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 Τέλος. Απορρίπτεται. Παράγραφος 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε για το τροποποιημένο κείμενο. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Ομόφωνα. Πέρασε. Μπράβο. Oh, It Ίσως είναι και η πρώτη φορά. Όχι, δεν είναι πρώτη φορά. Είναι σπάνιο πάντως, σπάνιο τόσο μεγάλη έκθεση, τόσο πολλές τροπολογίες είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να δούμε αν και ο Τσάλ θα μπορέσει να περάσει ομόφωνα τη δική του. Και η άλλη έκθεση ήταν πολύ σημαντική και περίπλοκο το θέμα. Ξεκινάμε λοιπόν πριν ψηφίσουμε, Σαρλ, στο 12 είμαστε της ημερήσιας διάταξης, η βιωσιμότητα του χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών. Σαρλ, θέλεις να πάρεις το λόγο. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές. Ελέγχουμε την 46. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος, απορρίπτεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος 47. Είστε υπέρ. Τέλος της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την 50. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 τα δύο τμήματα. Το πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Οι δύο άλλες αποσύρθηκαν. 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Όχι, όχι. Ελέγχουμε την 57. Όχι. 59. Όχι, όχι, όχι, όχι. Ελέγχουμε την 57. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 57. Τέλος. Απορρίπτεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 60 υπέρ. Το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται το 62. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 64. Τέλος. Εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εγκρίθηκε η 63. Πάμε στην 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66. Όχι. 67. 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να ελέγξουμε την 67. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 70 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ. Κατά αποχές. 71 ελέγχουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται. 72 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ. Όχι, 75 υπέρ κατά αποχές. Ελέγχουμε την 75. Τέλος. Απορρίπτεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την 77. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 79 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Για την 80. Τέλος. Απορρίπτεται. 81 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά αποχές, έλεγχος, 83. Ψηφίσατε όλοι, τέλος, εγκρίνεται. 85 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 86 υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε την 86. Μάλλον εγκρίνεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Προφορική 1. Υπέρ κατά. Απόχες. Έλεγχος για την προφορική 1. Τέλος. Εγκρίνεται. 89. Υπέρ κατά αποχές μάλλον απορρίπτεται ελέγχουμε την 89 ε, τέλος απορρίπτεται και τώρα περνάμε στην 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μπορούμε να την ελέγξουμε 90 Ελέγχουμε την 90. Τέλος. Εγκρίνεται. 91 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ. 95 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 96 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. 4. Ψηφίσατε όλοι τέλος. Εγκρίνεται. Πάμε στην 100 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2 προφορική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 104 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 109, όχι, όχι, όχι, 108, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 109 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 110 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 111 υπέρ, Α, ελέγχουμε την 110. Αρχή της ψηφοφορίας. Για την 110, τέλος, απορρίπτεται. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 112. Κατά. Πίπτη. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 114 υπέρ. 113. Απορρίφθηκε. Άρα πάμε στην 114, αφού απορρίφθηκε η 13. 114 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 116 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος 117. Ψηφίσατε. Τέλος. Καταπίπτει. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 118 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 118. Μάλλον εγκρίνεται. Τέλος. Εγκρίνεται. 119. Τα δύο τμήματα. Το πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 121. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 122 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε την 122 αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε. Τέλος. Απορρίπτεται. 123 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 124 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε την 125 ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. Είχατε δίκιο. Νομίζω ότι ήταν υπέρ απορρίπτεται 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 127 υπέρ κατά αποχές έλεγχος 127 αρχή της ψηφοφορίας τέλος απορρίπτεται 128 υπέρ κατά αποχές Έλεγχος 128. Ψηφίσατε, τέλος. Εγκρίνεται. 129 υπέρ. Κατά. Υπέρ, υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πάμε στην τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 5 αρχή της ψηφοφορίας ψηφίσατε όλοι τέλος εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ α συγγνώμη 8 8 υπέρ κατά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 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ. 20 υπέρ, κατά, αποχές. Ελέγχουμε την 20. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την 21. Μάλλον εγκρίνεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος για την 22. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. 23 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, ελέγχουμε την 26. Αρχή της ψηφοφορίας, 26, τέλος, εγκρίνεται. 27, όχι, 28, τα δύο τμήματα, το πρώτο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τελευταία σελίδα. 33 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 39 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 40 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο του κειμένου όπως έχει τροποποιηθεί. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίζουμε το τελικό κείμενο. Ψήφισαν όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Γκέρενς. Σας ευχαριστώ πολύ. 13 ψήφοι Ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες, συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τον πρόεδρο του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος θα πάρει το λόγο, θα μιλήσει για την κατάσταση στη Συρία. Όποιος θέλει να φύγει παρακαλώ πολύ ήσυχα. Συνάδελφοι, μπορούμε να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε ένα σημαντικό σημείο. Το σημείο 13. Αν σας παρακαλώ να καθίσετε, ε, θα δούμε το θέμα της κάλυψης ανθρωπιστικών αναγκών, η πρόκληση των παρατεταμένων κρίσεων. Χαίρομαι πάρα πολύ σήμερα, γιατί θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων με τον Πίτερ Μάουρερ, που είναι ο πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού από το 2012. Ελβετός, ο κ. Μάουρερ διετέλεσε υφυπουργός εξωτερικών της Ελβετίας στο παρελθόν, αλλά και περέσβης και μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελβετίας στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Μάουρερ Κύριε Μάουρερ, μάλλον είναι μεγάλη τιμή μας που σας έχουμε μαζί μας σήμερα. Ξέρουμε ότι η οργάνωσή σας έχει μακρά ιστορία, ιδρύθηκε το 1863 ως ουδέτερος οργανισμός με έδρα τη Γενέβη. Η ε, ο Ερθρός Σταυρός ε, ξεκινάει από τις συμβάσεις της Γενέβης του 1949. Ξέρουμε ότι ε, χειρίζεστε πολύ δύσκολες περιοχές του κόσμου και εσείς ο ίδιος επιστρέψατε τώρα από τη Συρία και το Ιράκ, πολύ δύσκολες χώρες. Ε, η χρηματοδότηση προέρχεται κυρίως από εθελοντικές δωρεές, από κυβερνήσεις και από τις εθνικές εταιρείες Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελίνου. Κύριε Μάουρε, έχω πολλές σημειώσεις, αλλά καλύτερα να μιλήσετε εσείς παρά εγώ για το έργο της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού, έναν οργανισμό τον οποίο στηρίζω στεναρά και όπως είπα, ε, ο οποίος λειτουργεί σε πολύ δύσκολες περιοχές με παρατεταμένες συγκρούσεις. Έχετε το λόγο λοιπόν κύριε Μάουραρ. Παρακαλώ ε, να παρακολουθήσουμε τον ομιλητή μας, τον κύριο Μάουραρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ που με φιλοξενείτε στην Επιτροπή σας σήμερα. Που μου δίνετε η δυνατότητα και η ευκαιρία να σας ενημερώσω για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, κάποιες από τις προκλήσεις. Ε, καθώς είμαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, ευχαριστήσω όλους εσάς για τη στήριξη, τη γενναιόδερη στήριξη στο έργο ε, της ΔΕΕΣ από τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, από την ΕΚΟ, από την ε, Επιτροπή εδώ στις Βρυξέλλες. Και αν βάλω όλα τα νούμερα μαζί, οι συνεισφορές οι ευρωπαϊκές στις εργασίες του ICRC είναι στα 47% ε, του προϋπολογισμού μας. Ε, και εδώ συμπεριλαμβάνονται κράτη-μέλη, ΕΚΟ ε, και θα ήθελα να δάξω την ευκαιρία να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα όλους εσάς για αυτή την πολύ γενναιόδερη στήριξη. Χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή να ανταποκρινόμαστε, να βοηθούμε ανθρώπους που έχουν ανάγκη ε, στην πρώτη γραμμή ε, των μαχών. Αντιλαμβάνομαι ε, και θα κάνω κάποια σχόλια στο δεύτερο ίσως μέρος της παρουσίασης, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι ε, μια από τις συζητήσεις σας εδώ στο Κοινοβούλιο και στις διαφορετικές επιτροπές είναι για το πώς ε, οργανώνετε την ε, οικονομική δομή έτσι ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να στηρίζετε την αναπτυξιακή συνεργασία, το ανθρωπιστικό έργο στο μέλλον. Υπάρχει μια συζήτηση που συνεχίζεται στη, σε αυτό το θέμα για τον καλύτερο τρόπο στήριξης αυτή τη διασύνδεσης ανάμεσα ε, στο ανθρωπιστικό και το αναπτυξιακό έργο με πιο, το, πιο αποτελεσματικό τρόπο. Θα ήθελα να αρχίσω ίσως με κάποιες από τις προκλήσεις που εμείς αντιμετωπίζουμε επί τόπου και πρόεδρε, αναφερθήκατε στις ε, πρόσφατες επισκέψεις μου στη Μέση Ανατολή, στο Ιράκ, στη Συρία. Ε, να σας δώσω μια σύντομη ανασκόπηση. Πάνω από 40% του έργου μας ε, συγκεντρώνεται στην Αφρική. Αφρική δηλαδή ε, τα καυτά σημεία συγκρούσεων που είναι το Σουδάν, η Σομαλία, η Λεκάνη, το λεκανοπέδιο της λίμνης του Τσάντ, ε, δηλαδή Νίγηρας, Καμερούν, Νιγηρία ε, και το Τσάντ. Εδώ είναι κατά δεύτερη σειρά μεγαλύτερες επιχειρήσεις μας, το Σαχέλ, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Εκεί έχουμε παρατεταμένες συγκρούσεις και εκεί ε, σε αναπτυξιακό επίπεδο και σε επίπεδο βίας ε, και συγκρούσεων έχουμε ε, προκλήσεις. Προκλήσεις που περιλαμβάνουν το πώς θα ε, πώς, ε, ε, λειτουργούμε και με άλλους φορείς, με άλλους οργανισμούς επιτόπου. Αν κοιτάξουμε τα τελευταία 7 χρόνια, η μεγάλη αύξηση του προπολογισμού του οργανισμού μας ήταν στη Μέση Ανατολή. Εκεί ε, ήταν μια περιοχή που δεν είχε δραστηριότητα ο Διεθνής Ερθρός Σαυρός, αλλά ο διπλασιασμός του του προπολογισμού μας τα τελευταία 7 χρόνια ε, έγινε ε, για τη Μέση Ανατολή. Τέσσερις από τις πέντε μεγαλύτερες επιχειρήσεις μας βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, μεγαλύτερη στη Συρία. Στη συνέχεια ακολουθεί ε, το Νότιο Σουδάν, η Εμένη, το Ιράκ, το Αφγανιστάν που είναι μεγάλα πεδία επιχειρήσεων ε, και προκλήσεων για μας. Τώρα, αν δούμε τις κυριότερες προκλήσεις, ποιες είναι αυτές, θα λέγαμε δύο μεγάλα κεφάλαια μας ανησυχούν. Πρώτον, η δυσκολία διαπραγμάτευσης πρόσβασης ε, σε έναν ε, ανθρωπιστικό χώρο. Πρόσβαση και ασφάλεια για τους εργαζόμενούς μας και πρόσβαση προς τον άμαχο πληθυσμό. Μπορώ να σας πω ότι ένα από τα μεγαλύτερα διλήμματά μου καθημερινά είναι σε ποιο βαθμό μπορούμε να πιέσουμε για πρόσβαση για να έχουμε ε, δέως επιμέλεια για το προσωπικό που επιχειρεί επιτόπου. Ε, δεν υπάρχει μαθηματικός τύπος για να το βρούμε αυτό, αλλά μπορώ να σας πω ότι ε, πιέζουμε όσο μπορούμε ως οργανισμός ε, η ατζέντα διαπραγμάτευσης πρόσβασης για να έχουμε πρόσβαση σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη επιτόπου στις χώρες αυτές όπου έχει διαταραχθεί εντελώς το κοινωνικό σύστημα. Είναι αυτό που κάνουμε στις περισσότερες ζώνες συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και αυτό έχει σχέση με την πρόκληση ε, ε, ότι το περιβάλλον είναι πολύ κατακαιρματισμένο. Ε, η Συρία και η Ιράκ δεν είναι ένα, ε, ε, ένα μέτωπο, είναι πολλαπλά μέτωπα, ίσως δεκάδες, εκατοντάδες παράγοντες που ενεργούν, με τους οποίους θα πρέπει να επικοινωνήσουμε έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ασφάλεια και ασφαλείς χώρους. Εάν πάμε στην Ανατολική Γούτα ή στη ε, Βόρεια Συρία ή σε κάποιες ζώνες του Αφγανιστάν, τότε εκεί υπάρχουν πολλαπλοί παράγοντες και φορείς με τους οποίους πρέπει να διαπραγματευτείς για να βρεις μια συνένεση, για να παρέχεις το ανθρωπιστικό έργο. Ε, πρόσβαση για ασφάλεια ε, στα μέτωπα είναι η πρωταρχική μας ανησυχία. Η δεύτερη ανησυχία, η δεύτερη πρόκληση που έχουμε και εδώ ε, είναι μια προκατάληψη που αντιμετωπίζω κάθε φορά που μιλάω ε, έξω από την ανθρωπιστική κοινότητα. Είναι ότι περισσότεροι θεωρούν το ανθρωπιστικό έργο ως έργο ανακουφιστικό, μετριασμού ε, των ελλημάτων της βίας, των προβλημάτων που προκαλούνται και των συνεπειών. Αλλά στην τελική ανάλυση η εντολή του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού είναι εντολή προστασίας Προσπαθούμε να έχουμε επαφή ε, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την, ε, την τήρηση του νόμου και την προστασία, γιατί ε, πρέπει να υπάρχει σεβασμός του διεθνού ανθρωπιστικού δικαίου. Υπάρχουν διαφορετικές πτυχές που μας απασχολούν σήμερα, βέβαια, στο θέμα αυτό. Πρέπει να έχουμε εμπλοκή με όλου, όλες τις δυνάμεις που ενεργούν επί τόπου σχετικά με την διεξαγωγή εχθροπραξιών. Προβλέπονται τρεις αρχές, προ, ε, αναλογικότητα, πρόληψη και ε, διάκριση ανάμεσα στους άμαχους και τους στρατιωτικούς. Και πρέπει να δούμε ε, ποιο είναι το νόημα αυτών των δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ανθρωπιστική μεταχείριση. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα για να διασφαλίσουμε ότι οι οικογένειες γνωρίζουν που βρίσκονται τα άτομα της οικογένειάς τους, των οποίο η τύχη αγνοείται. Και ε, ε, είναι ε, πράγματα που ήθελα να τονίσω. του, τους αριθμούς για τον προπολογισμό και η προσοχή συνήθως είναι στην πρόσβαση, στα, στην παροχή τροφίμων, και νερού σε περιοχές που είναι δύσβατες και δύσκολη πρόσβαση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά υπάρχει, ε, ε, υπάρχει και <clears throat> το θέμα ότι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε, αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές συνέπειες ε, του πολέμου αν δεν έχουμε μια ελάχιστη συμπεριφορά σε ό,τι αφορά τον σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Σήμερα θα έλεγα ότι υπάρχει ένα θέμα κάπου μεταξύ των προκλήσεων πρόσβασης και προσβασίας των ανθρώπων. Κάποιες είναι γύρω από θέματα υγείας, στήριξης ε, της υγείας και του τομέα της υγείας, τον οποίο ασχολούμαστε, διότι όλο ένα και πιο πολύ από αυτό που βλέπουμε από τη Συρία μέχρι το Αφγανιστάν και την Ιεμένη και σε πολλές άλλες περιοχές, είναι ότι η παράδοση ή απαγόρευση παράδοσης ε, υπηρεσιών υγείας είναι ένα από τα κρίσιμα ε, σημεία που προσπαθούμε να ξεπεράσουμε. Αν ε, εξετάσω τον χρόνο που διαπραγματευόμαστε στη Συρία, στο Ιράκ και ιδιαίτερα στην Ιεμένη και στη Συρία, που διαπραγματευόμαστε ένα πακέτο υπηρεσιών υγείας που να μπορέσουμε να το παραδώσουμε και που δεν παραδίδεται, από τις ε, δύο μεριές ε, των εχθροπραξιών είναι ένα δύσκολο θέμα. Έχουμε δυσκολίες ακόμα στο να ε, παραδώσουμε υλικό, ιατρικό, ιατροτεχνολογικό υλικό για χειρουργικές επεμβάσεις, γιατί πλευρές δεν μας επιτρέπουν να δώσουμε ανθρωπιστική βοήθεια στον τομέα της υγείας, ούτε ε, από ε, φάρμακα, ούτε από ε, υλικά, χειρουργικά υλικά. Επίσης, τα νοσοκομεία, τα συνοφόρα, τα σχολεία στοχεύονται κυρίως, είναι, αποτελούν στόχοι των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο αντίκτυπος ε, του πολέμου δεν επηρεάζει ατομικά τα άτομα, επηρεάζει τα συστήματα. Τι σημαίνει αυτό? Αν κοιτάξουμε την Ιεμένη και τη Συρία. Η Ιεμένη λειτουργεί στο ένα τρίτο της ε, υποδομής υγείας τώρα. Η Συρία στο 50% σε σύγκριση με την υποδομή προ του πολέμου. Δηλαδή 50% των νοσοκομείων και των κλινικών έχουν καταστραφεί ή υπολειτουργούν ε, αυτή τη στιγμή ή δεν λειτουργούν. 50% των γιατρών έχουν φύγει από τη χώρα, από τις χώρες, έχουν ε, σκοτωθεί, δεν ε, εργάζονται αυτή τη στιγμή εκεί. αυτή τη στιγμή που Υπάρχει μεγάλη πίεση για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ιδίως προς τους άμαχους που έχουν εμπλακεί ε, στη σύγκρουση. Ήθελα λοιπόν να αναφερθώ σε αυτά τα, αυτό τον σημαντικό πυλώνα δραστηριότητάς μας. Η πρόκληση επίσης είναι ότι οι συγκρούσεις είναι παρατεταμένες, όλα είναι και πιο πολύ, είναι μακροχρόνιες. Αυτή τη στιγμή έχουμε 30 χρόνια συν παρουσία στις 15 μεγαλύτερες επιχειρήσεις ε, μας ως διεθνής οργανισμός, δηλαδή ένας οργανισμός που δημιουργήθηκε για να παρέχει ε, βοήθεια έκτακτης ανάγκης, τώρα είναι για 30 χρόνια και στις μεγαλύτερες ε, επιχειρήσεις. Αυτοί οι αριθμοί αυξάνονται συνεχώς αυξάνονται ε, και, ε, αυξάνεται και η παράταση των συγκρούσεων και γίνονται και πιο περίπλοκες οι συγκρούσεις γιατί χαρακτηρίζονται από αστική βία, αστικές εχθροπραξίες, αστική σύραξη. Σημαίνει ότι είναι πιο τρωτή η υποδομή όταν μεταφέρεται ο πόλεμο στις πόλεις, ε, επηρεάζουν τα περισσότερα άτομα. Αν θέλετε να ξέρετε γιατί υπάρχει χολέρα στην Ιεμένη, αυτό σχετίζεται με τον πόλεμο. Ο πόλεμο έχει καταστρέψει τα συστήματα παροχή υδάτων ε, στι πόλει όπου ζουν οι άνθρωποι. Καταστρέφει τα νοσοκομεία και ένα συνδυασμό τη καταστροφή των συστημάτων υδατοπρομήθειας και νοσοκομείου σημαίνει ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο μία πόλη του ενός εκατομμυρίου δεν έχει ε, ούτε νερό ούτε συστήματα υγείας. Και ε, για, προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε τα συστήματα αυτά, αλλά πετυχαίνουμε το 80% το πολύ μετά την, ε, την πρώτη φάση του πολέμου. Αν υπάρχει δεύτερη φάση, ε, τότε είναι στο 50% η αποκατάσταση. Έχουμε συνεχή υποβάθμιση των συστημάτων υγείας, των συστημάτων υδατοπρομήθειας σε αστικό περιβάλλον γιατί η τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου σε ό,τι αφορά την αναλογικότητα και την διάκριση ε, δεν τηρείται. Εκεί όπου υπάρχουν οι εμπόλεμοι, οι αντίπαλοι που δεν τηρούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Αυτό που βλέπουμε, επίσης το ανάφερα και στην Αφρική, είναι η διασύνδεση της μακροχρόνιας φτώχειας μαζί με βία, με εγκληματική βία, με διακοινωτική βία, ενδοκοινωτική βία. Έχουμε ένα αρνητικό μείγμα που οδηγεί σε ένα πολύ ευθραυστό περιβάλλον που αποσταθεροποιεί ε, επίσης και το έργο της ανθρωπιστικής βοήθειας και ε, το σχεραίνει σε μεγάλο βαθμό. Ίσως να πω μερικά λόγια για το τι σημαίνει αυτό σε πολιτικό επίπεδο. Θα ήθελα να κάνω τρεις-τέσσερις παρατηρήσεις που υποθέτω και γνωρίζω ότι ε, απασχολούν ε, εσάς τους βουλευτές. Ένα θέμα το οποίο ε, οι βουλευτές συνήθως προβάλλουν είναι το πώς μπορείτε να δουλέψετε μαζί με άλλους και ποια είναι η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους αναπτυξιακούς φορείς και μακροχρόνιους ανθρωπιστικούς φορείς που ε, επιχειρούν σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. Θα προσπαθήσω να απαντήσω με τον εξής τρόπο. Εάν δούμε τις 20 μεγαλύτερες επιχειρήσεις μας σε παγκόσμια κλίμακα, που αποκλειστικά είναι ε, πλαίσια όπου υπάρχει μακροχρόνια βία και πόλεμος. Είναι τα κυρίαρχα στοιχεία που αντιμετωπίζουμε. Και υπάρχει και αμοιβαίο και αντιοτελές έργο λόγω της, ε, ότι υπάρχουν οι εμπόλεμοι ε, στο πεδίο της μάχης και υπάρχει η ανάγκη για διαπραγμάτευση ε, πρόσβασης. Αλλά δεν κάνουμε μόνο εκ τάκτο ανάγκη έργο ε, σε αυτές τις περιοχές, διότι είμαστε εκεί για 30 χρόνια και αντιμετωπίζουμε συνεχώ ένα νέο τύπο ανάγκης. Οι ανάγκες δεν είναι πια βράχυπρόθεσμες, είναι συστημικές και μακροπρόθεσμες. Και αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Τα κοινοβούλια και οι κυβερνήσεις δημιουργούν γραμμές προπολογισμού και διοίκηση που να αντιμετωπίζει το πρόβλημα, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει εξελιχθεί. Πριν από 30 χρόνια είχαμε αυτά τα αναπτυξιακά πλαίσια όπου η φτώχεια ήταν το κυρίαρχο θέμα και η μακροχρόνια αναπτυξιακή συνεργασία θα ήταν η καλύτερη αντιμετώπιση, ενώ είχαμε και βραχυπρόθεσμα προβλήματα εκτάκτου ανάγκης. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια ε, ανάμειξη, έχουμε μακροχρόνια συστημικό αντίκτυπο της βίας της κοινωνίας, όπου σημαίνει ότι η ανταπόκριση με μεθοδολογία ε, ε, πρέπει να αλλάξει, διότι ε, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε την ερεσιμότητα σε αυτό το πλαίσιο. Ένα άλλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση, δηλαδή πώς ε, τα κοινοβούλια μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτές τις καταστάσεις και να οργανώσουν τις αντίστοιχες υποδομές έτσι ώστε ως αναπτυξιακοί και ανθρωπιστικοί φορείς να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις. Και ειλικρινά μπορώ να σας πω ότι η καλύτερη λύση για μας θα είναι να υπάρχουν επαρκή κονδύλια σε, ανθρωπιστική γραμμή ε, προϋπολογισμού έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στα, ε, στις μεταβαλλόμενες ανάγκες με αμοιβαίο ε, και ανιδιοτελή τρόπο. Ε, αν δεν υπάρχει αυτή η επιλογή, τότε εμείς ενθαρρύνουμε πάντα τα αποθέματα τα οποία εσείς και οι άλλοι έχετε να ε, γίνονται διαθέσιμα για ε, την ανταπόκριση, την ανθρωπιστική που αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο. Και τρίτη λύση είναι να, υπάρχει να υπάρχουν ευελιξίες ανάμεσα στην στις ανθρωπιστικές και αναπτυξιακές γραμμές προπολογισμού πίστοσης που να μας επιτρέπει σε κάποιες περιπτώσεις να αντλούμε από αναπτυξιακά κονδύλια για να ανταποκριθούμε σε εύθραυστα πλαίσια, ιδιαίτερα σε μέρη όπου η έκτακτη ανταπόκριση ε, είναι για παράδειγμα για την επιδιόρθωση συστημάτων, όπου η έκτακτη ανταπόκριση μας δεν είναι απλά παράδοση τροφίμων σε εκτοπισθέντες, αλλά είναι στην ουσία να βοηθήσουμε τους αγρότες να ξαναρχίσουν τις δραστηριότητες τους και τη ζωή τους ε, μετά ή ε, και μέσα στη μέση της ε, σύγκρουσης. Θα ήθελα να σκεφτείτε δημιουργικά για την ε, διεπαφή της ανάπτυξης ε, και της, των ανθρωπιστικών προκλήσεων και να είστε όσο πιο ευέλικτοι μπορείτε, αλλά αναγνωρίζετε, αναγνωρίζετε πρέπει να είστε και να λογοθετείτε περισσότερο έτσι ώστε να προσαρμόζετε στην, αυτές τις αλλαγές που επιτελούνται σε ό,τι ε, στο τοπίο των αναγκών. Αυτό με ανησυχεί. Ε, γιατί πριν από 10 χρόνια θα ζωτούσατε τι, είναι ε, η ανθρωπιστική βοήθεια και θα σας έλεγε είναι ιατρική, είναι τρόφιμα, είναι στέγη, νερό. Σήμερα όταν ρωτώ τι σημαίνει και τι περιμένει κανείς από έναν ανθρωπιστικό φορέα, είναι η αποκατάσταση των σχολείων, είναι η έναρξη μικρών επιχειρήσεων και η στήριξη αυτών είναι η αποκατάσταση συστημάτων και επιδιόρθωση συστημάτων. Είναι ψυχοσωματική ε, ε, στήριξη για τραυματισμένα άτομα. Είναι στοιχεία ανταπόκρισης που πριν από 10 χρόνια δεν αποτελούσαν μέρος του κυρίως μέρους τη ε, της ανταπόκρισης της κρίσης. Ε, και ε, για το πώς ε, έπρεπε κανείς να ανταποκρίνεται. Θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να συζητήσουμε δημιουργικά για το πώς μπορούμε να βάλουμε τη, μια δομή οικονομική, διοικητική και λογοδοσίας έτσι ώστε να ανταποκρινόμαστε στις μεταβαλλόμενες ανάγκες σε αυτές τις ε, παρατεταμένες κρίσεις και συγκρούσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Ένα δεύτερο θέμα που σας ε, ανησυχεί πολιτικά είναι πώς η τα αναπτυξιακά και ανθρωπιστικά κονδύλια μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στη μετανάστευση ή μπορούν να έχουν σε ένα ε, βαθμό επίδραση στην πρόληψη της μετανάστευσης. Ένα μεγάλο θέμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε πολλές άλλες χώρες. Θα ήθελα και εδώ να επαναλάβω ότι είμαι υπέρ ε, ενός ανοιχτού και ε, επικριτικού διαλόγου ε, για τις πιέσεις που υφίστανται οι πολιτικοί στην Ευρώπη για το πότε είναι ασφαλές και σωστό να έχουμε θετική ανάπτυξη τα αναπτυξιακά κονδύλια και τα κονδύλια για τη μετανάστευση να χρησιμοποιηθούν για ανθρωπιστικούς σκοπούς. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Όταν βλέπω αυτά που έχω δει στη Συρία, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, Είμαστε υπερβολικά προσεκτικοί αυτή τη στιγμή για να συστήσουμε οποιοδήποτε, οποιαδήποτε μέσο, διευκόλυνση ή ενθάρρυνση επιστροφής πέραν από τον εθελοντισμό. Ε, ο καθένας θα πρέπει να καταλήξει στο δικό του συμπέρασμα και να κρίνει κατά πόσο νιώθει ασφαλής να επιστρέψει. Αλλά οποιαδήποτε ε, σχέδια εξαναγκασμένης επιστροφής αυτής της στιγμής, εκτός από ένα πολύ εύθραυστο πλαίσιο που βλέπουμε στη Συρία, στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, Πιστεύουμε ότι είναι πολύ πρόημο ακόμη το στάδιο για να γίνει αυτό. Στη Συρία είμαστε στη μέση μιας εκτάκτης ε, κρίσης και είναι απρόβλεπτο που θα καταλήξει η βία την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη μέρα. Στο Ιράκ έχουμε δει κάποιες θετικές εξέλιξεις μετά τη Μοσούλη, συμφωνώ, και υπάρχουν περιφέρειες όπου κάποιοι επιστρέφουν. Από τα 5 εκατομμύρια που εκτοπιστήκαν, 2,5 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένοι έχουν επιστρέψει στις αιστείες τους. Αλλά θα ήθελα να σας πω ότι 2,5 εκατομμύρια Ιρακινοί εξακολουθούν να είναι εκτοπισμένοι αυτή τη στιγμή και δεν μπορούν να επιστρέψουν γιατί οι υποδομές, ε, τα σπίτια έχουν καταστραφεί και οι απαραίτητες βασικές υποδομές βοήθειας για να ανοικοδομήσουν το περιβάλλον τους δεν υπάρχουν. Η πολιτικός είναι πρόημο να στείλουμε αυτούς τους ανθρώπους πίσω, διότι πολλές κοινότητες ακόμη είναι μικτές, ε, Σιά, Σούνις, Κούρδων, Αραβών και είναι ε, έντονα διχασμένοι, άρα υπάρχει ακόμη η βία ε, που απαιτεί προφύλαξη. Θα ήθελα όμως για άλλη μια φορά να πω ότι πρέπει να έχουμε ανοιχτό πνεύμα, ε, ένα ανοιχτό διάλογο. Δεν είναι όλα τα μέρη μη ασφαλή και δεν είναι πάντα αδύνατο να ενθαρρύνουμε έστω την εθελούσια επιστροφή και με την πάροδο του χρόνου να έχουμε ισχυρότερη ενθάρρυνση για αυτή την επιστροφή. Ένα τρίτο σύντομο σημείο που θέλω να θίξω είναι ότι σήμερα ακούμε συνεχώς για την τοπικοποίηση της ε, βοήθειας και ως μέλος της οικογένειας του Ερυθρού Τσαυρού και της Ερυθράς Εμισελίνου θα ήθελα να σας πω πόσο εκτιμούμε το έργο με τις ε, αντίστοιχες ε, εθνικές εταιρείες στις περιοχές που επιχειρούμε με την Ερυθρά Εμισιαλίνο της Συρίας και άλλες εταιρείες που συνεργαζόμαστε. Τούτου λεπτέντος όμως θα ήθελα να είμαι πολύ σαφής. Ε, σε μια, ένα από τα προβλήματα είναι ότι οι ντόπιοι είναι μέρος της σύγκρουσης και του προβλήματος στη χώρα και η ανάπτυξη αμοιβαία ανταπόκρισης ανθρωποστικής όταν η χώρα είναι ακόμη στη μέση μιας σύγκρουσης και όταν το προσωπικό σου και το εθνικό προσωπικό ε, είναι μέρος της σύγκρουσης περισσότερο από το διεθνές προσωπικό, αυτό αποτελεί συνταγή για αποτυχία. Εγώ αυτό το οποίο υποστηρίζω είναι και πάλι να έχουμε μια πιο έξυπνη χρήση και αλληλεπίδραση ανάμεσα στους διεθνείς και τους εθνικούς φορείς ε, ανταπόκρισης. Σήμερα η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού είναι η καλύτερη εταιρεία διασφάλισης για τον, την ημισέλινο στη Συρία που είναι ε, ε, αυτή τη στιγμή αν μείνει μόνη της είναι πολύ τρωτή στις επιθέσεις διότι είναι μέρος της κοινωνίας και του ιστού της κοινωνίας και δεν είναι τυχαίο που η Μισέλινος στη Συρία έχει τα περισσότερα θύματα σε αυτή την σύγκρουση στη Συρία. Άρα εγώ θα ακολούθησα το παράδειγμα και θα το πρότεινα να το μελετήσετε, να, έχουν, να δούμε πού ε, ένας διεθνής φορέας θα μπορούσε να διαδραματίσει ένα ρόλο, ιδιαίτερα σε ε, παρατεταμένες συγκρούσεις, όπου οι ντόπιοι μπορούν να έχουν καλύτερο τρόπο να βρουν τρόπο ανταπόκρισης. Και τέλος, όπως και πολλοί άλλοι φορείς σήμερα και εμείς, σκεφτόμαστε και μελατούμε για το πώς μπορούμε να διαφοροποιήσουμε ε, και να καινοτομήσουμε ε, στους τρόπους ανταπόκρισης μας, η ψηφιοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, η διασυνδεσιμότητα που μας συνδέει με διαφορετικούς τρόπους με τους ε, με, με αυτούς που επωφελούνται επί τόπου αλλάζει τον τρόπο ανταπόκρισης και θα πρέπει να διαρευνηθεί αυτό. Θα πρέπει να το δούμε, να το εξετάσουμε, να το μελετήσουμε και το κάνουμε. Φέτος ε, δεν έχουμε μόνο να διαμορφώσει την θεσμική μας στρατηγική, αλλά και την ψηφιακή μας στρατηγική. Ελπίζουμε ότι θα μας καταστήσει ε, κορυφαίους ε, στην ανταπόκριση, χρησιμοποιώντας τον κυβερνοχώρο, έτσι ώστε να επιτελούμε καλύτερο ανθρωπιστικό έργο. Και αυτό από, ξεκινώντας από ένα ασφαλές αποθετήριο ε, δεδομένων μέχρι και τη χρήση δεδομένων για να παρέχουμε ανθρωπιστική βοήθεια και σε άλλα θέματα τα οποία επίσης μελετούμε. Έχουμε ακρηγορήσει, αλλά ήθελα να σας δώσω μια εισαγωγική εικόνα για τις ε, ανησυχίες μας σήμερα. Ευχαριστώ. No, I think it's Νομίζω ότι είναι σημαντικό. Δεν έχουμε πάντα τον πρόεδρο του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού εδώ, επομένως ε, είναι σημαντικό να σας δώσουμε χρόνο να μας μιλήσετε για το έργο σας. Ε, να σας πω ότι όλα αυτά τα θέματα που αφορούν ε, το, την ευρασία και την ψηφιοποίηση μας απασχολούν και μάλιστα σήμερα συμφωνήσαμε για μια έκθεση για την ψηφιοποίηση και την βοήθεια. Ίσως λοιπόν θα μπορούσατε να μας τροφοδοτήσετε κι εσείς μέσω του γραφείου σας η ομάδα του ΕΛΚ θα ορίσει ε, αρμόδιο εισηγητή για την ψηφιοποίηση και για την χρηματοδότηση και την οργάνωση της χρηματοδότησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά μια διαδικασία αναθεώρησης όλων των κονδυλίων για το θεματολόγιο του 2030 και ε, τα προγράμματα από το 2020 και μετά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το πώς θα, είναι, ε, πώς θα εφαρμοστούν στην πράξη Τώρα λοιπόν είναι η κατάλληλη στιγμή να τα δούμε όλα αυτά. Μας απασχολούν όλα αυτά τα θέματα. Ευπρόσδεκτες λοιπόν και ε, οι δικέ σα οι απόψει και η συμβολή σα στο θέμα αυτό. Ο Σαλ Κέρενς θέλει να ξεκινήσει. Παρακαλώ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Μωρέ, τον πρόεδρο της, ε, τον πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού. Ξέρουμε σε ποιο βαθμό ασχολείστε με ανθρωπιστικά ζητήματα και φυσικά δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσουν αυτά που κάνετε. Κάποιες ερωτήσεις. Πρώτον, η οργάνωση από πλευράς Γενέβης. Είστε πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και υπάρχει και η Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού, τη διεθνή Ομοσπονδία των Εθνικών Ερυθρών Σταυρών. Σε ποιο πλαίσιο προβλέπετε να παρεμβάνει η μία ή η άλλη οργάνωση. Νομίζω ότι γνωρίζω, αλλά καλό θα ήταν ε, να μας το υπενθυμίσετε και εδώ. Δεύτερο, το έγγραφο Responsibility to Protect. Ξέρουμε ότι ένας ε, εκ των προκατόχων σας είναι ο ένας από τους συντάκτες αυτού του εγγράφου και το έγγραφο αυτό προβλέπει και την υποχρέωση προστασίας, ε, παροχής ασφάλειας και κατά την άποψή μου αυτό πηγαίνει λίγο πέραν ε, της ουδέτερης και αμερόληπτης εντολής της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού. συμφωνείτε απολύτως με τις ε, συστάσεις αυτού του εγγράφου ή ο κύριος Αμπρούγκα παρουσιάζει τις προσωπικές του απόψεις, διότι όταν συνέταξε το κείμενο δεν ήταν πλέον πρόεδρος της ε, Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού. Είσαι Σιλκιέγγε, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και εγώ για την ε, συμβολή σας εδώ και θα ήθελα να πάρω το λόγο για τρία θέματα. Πρώτον, αναφερθήκατε στην διαφοροποίηση της ε, χρηματικής βοήθειας. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει σύγκληση των διαφέρων μέσων χρηματοδότησης ε, και στην ε, βοήθεια, διότι σε πολλές από αυτές τις περιοχές κρίσης και σύραξης η βοήθεια για την ανάπτυξη θα πρέπει να είναι περιορισμένη χρονικά, αλλά πρωτίστως πρέπει να βοηθά τα μέσα που υπάρχουν επιτόπου να είναι καταλήτης, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ανθεκτικότητα, να δώσουμε στα χέρια των ανθρώπων επιτόπου τη δυνατότητα να μπορούν να πάνε πέραν της λογικής, της βοήθειας, διότι τη στιγμή που θα τελειώσει η βοήθεια, οι άνθρωποι αυτοί είναι εξαρτημένοι πλέον και είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσουν να προχωρούν. Η διαφοροποίηση λοιπόν των διάφορων μέσων και η σύγκλησή τους θα πρέπει να ενισχύσει αυτό που συζητούμε σήμερα, την ανθεκτικότητα, να προσφέρουμε αυτονομία και δυνατότητα στις διάφορες περιοχές να προχωρήσουν. Ε, το δεύτερο είναι ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται στη χρήση και στη διαχείριση της βοήθειας. Ε, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ανθρωπιστικές οργανώσεις, αλλά πολύ συχνά υπάρχει συμμετοχή και τοπικών φορέων. Θα αναφερθώ σε δύο περιπτώσεις, αλλά θα μπορούσα να επεκταθώ και σε άλλες. Η περίπτωση της λαϊκής δημοκρατίας του Κονγκό, ε, στην οποία αυτή τη στιγμή υπάρχει ε, κρίση ασφάλειας, ε, πολιτική και ανθρωπιστική, πολύ βαθιά. Και αν περάσει κάποιος από τις κυβερνητικές ή θεσμικές αρχές, εγώ θεωρώ τρόπον την ότι δίνουμε, ε, αυτό αποτελεί κόλαφο για το λαό, διότι είναι υποκαθεστώς καταπίεσης και αυτό είναι από τον κυβερνητικό μηχανισμό εντός των θεσμών. Υπάρχουν έρευνες εν εξελίξη ήδη αυτή τη στιγμή για ε, ε, προσώπους των Ηνωμένων Οθνών που σκοτώθηκαν ε, και υπάρχουν υποψίες ότι οι δολοφονίες ήταν έργο των ίδιων των κυβερνητικών θεσμών. Και πραγματικά αυτή η βοήθεια φτάνει επί τόπου και πηγαίνει στα χέρια ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι για τη δολοφονία και την καταπίεση πολλών ανθρώπων. Τι άποψη έχετε εσείς επ' αυτού. Και το ίδιο θα μπορούσα να το πω και για μια χώρα όπως το ε, Μάλι, στο οποίο η κατάσταση είναι καταστροφική. Πριν από μια εβδομάδα ήμουν στο Μάλι και διαπίστωσα, η δύσομασία, ότι η κατάσταση είναι τόσο δραματική που αν δεν κάνουμε κάτι στο επόμενο εξάμεινο θα βρεθούμε αντιμέτωποι με μία ακόμα κρίση, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει, διότι να σας υπενθυμίσω ότι ε, η Μινούσμα είναι μία από τις δυνόμεις που έχασε και είχε τις μεγαλύτερες ε, ανθρώπινες απώλειες ε, από όλε τι ε, ειρηνευτικέ δυνάμει. Ε, και λοιπόν η Λαϊκή Δημοκρατία και το Μάλι, ε, του Κονγκό και το Μάλι έχουν το ίδιο πρόβλημα. Πώς μπορούμε να περάσουμε από τι κυβερνητικέ δομέ, γιατί δεν ξέρουμε και σε ποιον να αποτανθούμε σε αυτή την περίπτωση. Ε, τρίτον, η προστασία των ανθρώπων. Ε, είδαμε ότι κάποιοι οποίοι πήγαιναν να προσφέρουν βοήθεια στο Αφγανιστάν από το Save the Children ε, επιθέσει επιθέσεις πριν από μερικές εβδομάδες. Και βλέπω ότι οι άνθρωποι που πηγαίνουν να προσφέρουν βοήθεια ε, όλο ένα και αραιώνουν. Ε, μπορείτε να μου πείτε και εσείς την άποψή σας, διότι το να πάει κάποιος σε μια περιοχή σύγκρουσης και εδώ να επανέλθω και στη δολοφονία των δύο αποσταλμένων των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίοι δολοφονήθηκαν στο Κασάι, γιατί ε, στάλησαν σε μια περιοχή ε, με πολύ μεγάλο κίνδυνο, χωρίς καμία προστασία. Η μία εξ αυτών ήταν μια Σουηδή και ο άλλος ήταν κάποιος... Ε, από τις Ηνωμένε Πολιτείες. Θα ήθελα να ξέρω τι άποψη έχετε εσείς για τους ανθρώπους οι οποίοι μεταβαίνουν σε περιοχές ε, ανοιχτή σύγκρουσης και κρίσης ε, ε, ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο. Έχω τον Ερίκε Γκερέρο που χρειάστηκε να φύγει γιατί είχε μια συνεδρίαση στις 12 και αναχώρησε, ζητά συγγνώμη που δεν μπόρεσε να παραμείνει και ήθελε να υποστηρίξει αυτά που είπατε για την προσφορά. Δεν ε, μπορούμε να προσφέρουμε απλώς ε, μόνο ψυχολογική υποστήριξη στους ανθρώπους που βρίσκονται σε περιοχές σύγκρουσης, αλλά χρειάζονται περισσότεροι ιατρικές ε, ανάγκες και είδαμε επιτόπου, διότι εγώ Πήγα στο δόκτωρ ε, Μακουίγκη στο νοσοκομείο του στο Πάντζι πριν από κάνα δύο χρόνια με τη Σεσίλ Κέγγε και είδαμε ε, επιτόπου τι προβλήματα υπάρχουν και τι περιορισμοί στην ανθρωπιστική βοήθεια. Για παράδειγμα, του δόθηκαν χρήματα για να βοηθήσει οι γυναίκε που είναι θύματα βία, αλλά ζει σε μια περιοχή ε, απόλυτη φτώχεια και μια γυναίκα έρθει λοιπόν στο νοσοκομείο απλώ γιατί είχε πρόβλημα κατά τη γέννα με το παιδί τη. Δεν είναι μόνο πρόβλημα βία, αλλά είναι πάρα πολύ φτωχή. Ε, δεν μπορεί να κάνει τέτοια διάκριση όταν ε, προσφέρει θεραπεία σε αυτές τις γυναίκες και είναι λίγο θολά τα όρια σε αυτές τις περιοχές. Και την όλη συζήτηση που θα κάνουμε για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και τα νέα προγράμματα, κάτι το οποίο είναι συχνά χρήσιμο, είναι αντί να μας παρουσιάζεται το πρόβλημα σε θεωρητικό επίπεδο, όπως κάνουμε συνήθως ε, στον ε, κόσμο της αναπτυξιακής βοήθειας, ε, είναι πολύ πιο εύκολο να αντιληφθούμε απτά προβλήματα, να περιγράψουμε ότι στην τάδε περιοχή θέλαμε να κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό γιατί, και δεν μπορούσαμε να το κάνουμε γιατί δεν δόθηκε η κατάλληλη βοήθεια. Έτσι ο κόσμος αντιλαμβάνεται πολύ πιο εύκολα την πραγματικότητα των περιορισμών που υπάρχουν στη χρηματοδότηση. Για παράδειγμα, πήγαμε επί τόπου σε μια χώρα και είδαμε ότι δίνονται χρήματα για να εκπαιδευτεί ο στρατός από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουν να ε, αναλάβουν τα ενία και να πάρουν τον έλεγχο από ένοπλε ομάδε. Και καταλάβαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να βοηθήσει. Ναι, μεν εκπαιδεύουμε το στρατό, αλλά η χρηματοδότησή μα δεν μπορεί να βοηθήσει, δεν μπορούν να του δώσουν στολέ, για παράδειγμα. Το πρόβλημα γίνεται πολύ πιο ε, διαφορετικό και υπαρκτό αν μα δώσετε συγκεκριμένα παραδείγματα, αν έχετε συγκεκριμένα αυτά παραδείγματα πραγμάτων που είδατε επί τόπου, αυτό θα μπορέσει να μα βοηθήσει να αντιληφθούμε και τη φύση των προβλημάτων. Πριν λοιπόν να σας ξαναδώσω το λόγο για να απαντήσετε σε ερωτήσεις, νομίζω ότι έχουμε εδώ εκπροσώπου της Γενικής Διεύθυνσης ΕΚΟ. Να μας συστηθείτε γιατί δεν βρίσκω το όνομά σας στον κατάλογο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Λέγομαι Πατρίς Λενογμό και είμαι στην μονάδα Eco Strategic Unit. Πολύ σύντομα Τρία σημεία. Θέλω καταρχήν να πω ότι εννοείται ότι ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός είναι ένας από τους πιο σημαντικούς εταίρους που έχουμε σε πολλές περιοχές, Ουκρανία, Αφγανιστάν, Μέση Ανατολή. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καμία πρόσβαση χωρίς εκείνους. Σημαντικότατη λοιπόν συνεργασία και εταιρική σχέση. Όπως είπε ο πρόεδρος Μόρελ για θέματα ανθρωπιστικού δικαίου, προστασία συνόρων. Αυτό είναι προτεραιότητα για μας και βεβαίως συνεχίζουμε να δραστηριοποιούμαστε όπως μπορούμε και στη Συρία. Για άλλη μια φορά η βοήθεια και η στήριξη του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού είναι σημαντικό. Σήμερα έχουμε ομήρους, έξι που δολοφονήθηκαν στην περιοχή αυτή και δυστυχώς ένα μεγάλο τμήμα αυτών των ομήρων και αυτών που πλήττονται και δολοφονούνται είναι μέλη του Διεθνούς Ευθυνού Σταυρού. Ο Σάρλ θέλει πάλι το λόγο. Να προσθέσω μια άλλη ερώτηση σε αυτή που μόλις έκανα. Ξέρω ότι είναι αμερόληπτη η οργανωσή σας, ο Ερυθρός ε, Σταυρός τι πιστεύετε για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά την υιοθέτηση αυτού του Global Act και πώς εσείς μπορείτε να συνεχίσετε τις δραστηριότητές σας επιτόπου από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί πλέον η πολυμερής παρέμβαση σίγουρα σας εμποδίζει σε περιοχές με σύγκρουση να δραστηριοποιηθείτε, να είστε αποτελεσματικοί. Για μας αυτό είναι απαράδεκτο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να βρει λύσεις, να συνεχίσει να συνεργάζεται πιο στενά μαζί σας έτσι ώστε οι αρνητικές συνέπειες αυτού του καταστροφικού νόμου να αντιμετωπιστούν. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω με την ερώτησή σας. Αυτό που εμείς προτείνουμε είναι να μην αντιμετωπίσουμε με θεωρητικό ή γραφειοκρατικό τρόπο αυτά τα πράγματα. Είμαστε επιτόπου, οι άνθρωποι εργάζονται στις περιοχές αυτές, δύσκολες περιοχές και καθημερινά προσπαθούμε να αξιολογήσουμε τις ανάγκες και να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία προκύπτουν. Δυστυχώς βλέπουμε ότι υπάρχει και η γραφειοκρατία και οι πιστώσεις στον προϋπολογισμό οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τις ανάγκες των ανθρώπων επιτόπου. και πολλές φορές υπάρχουν ανάγκες οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν άμεσα εάν θέλουμε να συνεχίσει η ζωή στις περιοχές αυτές. Και θα σας πω κάτι το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της δράσης μας, όπως και όλων των ανθρωπιστικών ε, οργανώσεων. Οι άνθρωποι βρίσκονται στην καρδιά της ανησυχίας μας και της δράσης μας. Ίσως θα σας φανεί λίγο ε, συνηθισμένο αυτό σαν φράση, αλλά πραγματικά κάθε στιγμή προσπαθούμε να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες. Ανάγκες που μεταβάλλονται, που αλλάζουν. Να βάλουμε στην καρδιά της ε, δράσης μας τους ανθρώπους και να προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε τις ε, ανάγκες τους. η γραφειοκρατία και οι γραμμές του προϋπολογισμού, η κάλυψη των αναγκών δηλαδή αυτών, κάνει μία ταξινόμηση των αναγκών. Οι ανάγκες ε, οι οποίες ε, ταξινομούνται ως ανθρωπιστικές, οι άλλες που ταξινομούνται ως ανάγκες σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Ε, αυτά όμως στην πράξη δεν υπάρχουν. Υπάρχουν ανάγκες ανθρώπων τις οποίες εμείς πρέπει να καλύψουμε. Και γι' αυτό το θέμα, αν θέλετε, των αναγκών των ανθρώπων θα πρέπει να βρίσκεται ολοκληρωτικά και ε, σε κάθε περίπτωση στο κέντρο των προτεραιοτήτων μας. Εάν ακούει κανείς τον κόσμο, τους ανθρώπους, σίγουρα θα είχαμε διαφορετικά προγράμματα εντελώς διαφορετικά προγράμματα ανθρωπιστικής δράσης. Για μας λοιπόν αυτό είναι το καθοριστικό πριν ε, δραστηριοποιηθούμε και πριν φτιάξουμε ένα πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα πρέπει να ξεκινάει από κάτω, bottom-up, να ξεκινάει από τις ανάγκες των ανθρώπων και να προσπαθούμε να χτίσουμε το κάθε σχέδιό μας, το κάθε πρόγραμμά μας βάσει αυτών. Και αυτό σίγουρα είναι κάτι λίγο πιο αξιόλογο από το να ταξινομεί κανείς τις ανάγκες των ανθρώπων. Χρειάζεται ευελιξία όσον αφορά τη χρηματοδότηση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις πραγματικές ανάγκες στην δράση. Ε, στην πράξη βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ μικρές επιχειρήσεις, πολύ μικρές, ε, πολύ ε, οργανισμοί, φορείς ε, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη δράση και συνεργάζονται μαζί μας. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα και πώς εξοπλίζουμε την δική μας οργάνωση για να μπορέσουν να είναι αποτελεσματικοί στην πράξη. Η οργάνωσή μας, ο Διεθνής Ερυθρό Σταυρό είναι μία μικιό ελβετική. Αυτό είναι το καθεστώς μας. Και η Ελβετική Ομοσπονδία συντονίζει από εκεί συντονίζεται η δράση μας για φυσικές καταστροφές και κάθε άλλου είδους περιπτώσεις όπου παρεμβαίνουμε από εκεί ενδεχομένως ξεκινάει το πρόβλημα. Σήμερα το περιβάλλον είναι εξαιρετικά περίπλοκο και υπάρχει η σύγκρουση, η βία και τα κοινωνικά προβλήματα τα οποία καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε. Και βεβαίως καλούμεθα να ανταποκριθούμε σε όλες αυτές τις προκλήσεις. 15-20 εξαιρετικά βίες συγκρούσεις τις οποίες παρεμβαίνουμε. Είμαστε συντονιστές της δράσης επιτόπου με τον, την Τράι ε, Σέλινο και άλλους οργανισμούς και θα βεβαίως να κάνουμε αυτό που είναι αν θέλετε η καρδιά της δράσης μας αλλά όχι μόνο σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Η Ομοσπονδία είναι αυτή που αναλαμβάνει τη δράση και κάνει το συντονισμό. Η Ομοσπονδία του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Θα ήθελα επίσης να απαντήσω στην ερώτηση που αφορά την ανθρωπιστική δράση, λέγοντας ότι ναι, πρόκειται για μια δράση που σίγουρα είναι συνενετική καταρχήν. Γι' αυτό και κάθε φορά σαν ε, θεσμός προσπαθούμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Παραδείγματος χάρη, υπό την ε, σύμβαση της ε, Γενέβης, πολλές φορές η δράση μας ε, φτάνει σε κάποια αδιέξοδα. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της συνένεσης και το θέμα της εθνικής ε, κυριαρχίας παραδείγματος χάρη, το οποίο πολλές φορές δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε, ακόμα και αν επικαλούμαστε την υποχρέωση που έχουμε να παρέμβουμε και να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή. Ο Κορνέλιος Ομαρούγκα που βεβαίως και όταν έπαψε να είναι πρόεδρος του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, συμμετείχε στη σκέψη γύρω από όλα αυτά τα θέματα και αν θέλετε αφιέρωσε δύο χρόνια ε, τη ζωή του για το θέμα αυτό της ανθρωπιστικής δράσης, λέγοντας ότι δεν αρκεί το ότι είναι συνενετική αυτή η δράση. Πολλές φορές περιορίζουμε τη δράση μας για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να δρούμε με ουδετερότητα, με αμεροληψία, και να βασιζόμαστε σε μια συνενετική υποστήριξη. Όσον αφορά την ερώτηση που αφορά τους τοπικούς φορείς και οργανισμούς, όπως και η Εθνική Ερυθρή Σταυρή ανά τον κόσμο, όπως και οι άλλοι που δραστηριοποιούνται Μισέλινος, προσπαθούμε να είμαστε πολύ κοντά στις τοπικές κοινότητες. Από την άλλη πλευρά, όλοι αυτοί οι τοπικοί φορείς και οργανισμοί είναι πολύ πιο εύκολο να αποτελέσουν αντικείμενα χειρισμού από τις στρατιωτικές αρχές, τις πολιτικές αρχές και τις κυβερνήσεις επιτόπου. Άρα δεν υπάρχει ένας γενικός κανόνας ο οποίος εφαρμόζεται παντού. Κάθε φορά προσπαθούμε να αξιολογήσουμε με μεγάλη προσοχή και να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να προστατεύσουμε τοπικές πρωτοβουλίες από πιθανές καταχρήσεις. Έχουν πολλά πλεονεκτήματα οι τοπικοί φορείς και οργανισμοί γιατί είναι πολύ πιο κοντά στις τοπικές κοινότητες, αλλά και εμείς θα πρέπει να τους προστατεύσουμε από πιθανούς χειρισμούς, έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η δράση τους η κατάσταση, όπως είπατε, στο Κονγκό, ιδιαίτερα σε κάποιες περιοχές, είναι εξαιρετικά δύσκολη. Και εκεί προκύπτει και ένα άλλο δίλημα, προληπτική δράση. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά την προληπτική διπλωματική αποστολή που προσπαθούμε να αναπτύξουμε, γιατί οι διεθνείς υποδομή για αναπτυξιακή βοήθεια, για ανθρωπιστική βοήθεια, προϋποθέτει να υπάρχουν κάποιες τοπικές αρχές με τις οποίες να συνεργαστούμε. Σήμερα καταλαβαίνετε ότι το ανθρωπιστικό δίκαιο όταν έχεις απέναντί σου ένοπλες ε, ομάδες και καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, η δράση μας ε, βεβαίως είναι πάντα αδύναμη και δεν αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματα. Και εδώ επανέρχομαι στο θέμα των ε, χρηματοδοτικών ε, δυνατοτήτων. Χρειαζόμαστε διαφορετικά εργαλεία χρηματοδοτικά, αλλά και διαφορετικό τρόπο απάντησης και κάλυψης διαφορετικών αναγκών. Υπάρχει η στήριξη βάση των ε, αναπτυξιακών ε, στόχων αλλά και όλες αυτές οι προϋποθέσεις και οι όροι για να είναι αποτελεσματική η ανθρωπιστική βοήθεια. Είτε διαχειρίζεται κανείς τους πόρους αυτούς με έναν ολοκληρωμένο τρόπο ή το κάνει με διαφορετικό τρόπο, αυτό που είναι σημαντικό είναι να παραμείνει κανείς ουδέτερος, αμερόληπτος στην ανθρωπιστική στήριξη που προτείνει για να μπορέσει πραγματικά να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ανθρώπων αυτών που βρίσκονται σε δραματική κατάσταση. Δεν μπορεί μονίμως να χρησιμοποιούμε την ίδια μεθοδολογία και τους ίδιους τρόπους. Πρέπει να αποφεύγουμε επικαλύψεις, να βρούμε τρόπους να δημιουργήσουμε συμφιλίωση, να καθορίσουμε πολιτική που να προλαμβάνει τα προβλήματα, της δυσκολίες. Και πάνω απ' όλα θέλουμε να προστατεύσουμε τους ανθρώπους με ευελιξία. Χρειάζεται ευελιξία, χρειάζεται αλλαγή όσον αφορά την παρέμβαση και τη δράση μας. Και αυτά είναι βεβαίως πολύ σημαντικά προβλήματα και αδυναμίες που συνεχίζουμε να έχουμε. Και πολλές φορές βλέπουμε ότι εν μέσω σειράξεων και συγκρούσεων η κατάσταση δεν είναι ε, ευνοϊκή για την δική μας παρένθεση. Δεν είναι τυχαίο το ότι πέρσι στα πλαίσια της κρίσης στην Σομαλία η Εμένη μας πλησίασε η Παγκόσμια Τράπεζα. Συνεργαστήκαμε μαζί τους. Η Παγκόσμια Τράπεζα μπορεί να παρέχει κονδύλια σε κάποιες αναπτυξιακές υπηρεσίες, αλλά όσον αφορά τη σταθεροποίηση, όσον αφορά θέματα που αφορούν κρίσεις επιτόπου για άμεση αντιμετώπιση καταστροφών είτε της πείνας. Εμείς πρέπει πραγματικά πάντα να έχουμε κατά νου την ευελιξία που είναι απαραίτητη για να αποφύγουμε την ε, επικάλυψη και για να σιγουρευτούμε ότι τα χρήματα, η ανθρωπιστική βοήθεια πάνε πραγματικά σε αυτούς που τα έχουν περισσότερο ανάγκη. Αλλά σίγουρα κάθε φορά που υπάρχει μια τέτοιου είδους κρίση πρέπει να προσαρμόσουμε την ε, δράση μας. Uh, σχετικά με την προστασία των ανθρωπιστικών εργαζομένων είναι ένας εφιάλτης λόγω του κατεκερματισμού της ε, απρόβλεπτης φύσης των παιδιών μαχών. Μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν δύο φιλοσοφίες που ισχύουν. Πρώτον, αυτήν που την ενθαρρύνεται ο Διεθνής Ερθρός Σταυρός και είναι διαφορετική από το σύστημα του ΟΗΕ. Το σύστημα του ΟΗΕ προστατεύει ε, με όπλα και ειρνευτικές δυνάμεις και ε, διασφάλιση του ανθρωπιστικού έργου. Εμείς ε, δουλεύουμε με τις διαπραγματεύσεις και την οικοδόμηση συνένεσης. Δεν στηριζόμαστε στην ασφάλεια με τη χρήση των όπλων και αν δείτε το αποτέλεσμα, και οι δύο οργανισμοί έχουμε προκλήσεις σε ό,τι αφορά την διασφάλιση των επιχειρήσεών μας και τις λειτουργίες μας, αλλά δεν ισχύει ότι η χρήση όπλων ε, στο ανθρωπιστικό έργο μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη ασφάλεια για τους ανθρώπους επιτόπου. Το έργο οικοδόμηση συνένεση με τους κύριους παίκτες ε, στο πεδίο της μάχης είναι σίγουρα απαραίτητο και κρίσιμη σημασίας. Νομίζω έχω απαντήσει, ναι. Ε, οι διερμηνείς μπορούν να αποδεσμευτούν